Okay, chers collègues, je vous propose de commencer. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε, θα σας πρότεινα. Chers amis, j'ouvre la séance. Donc, on a... Ξεκινούμε λοιπόν ε, την ημέρα διάταξη, πρέπει πρώτα να την εγκρίνουμε βέβαια να πω για το θέμα αυτό ότι θα υπάρξει ένα αίτημα να αναβληθεί η ψηφοφορία ε, όχι τώρα όμως διότι δεν θέλω να χαθεί χρόνος γι' αυτό τώρα θα το δούμε την κατάλληλη στιγμή μπορείτε να ακούσετε όλες τις γλώσσες έξω από τα μαλτέζικα, τα κροατικά, τα φιλανδικά και τα σλοβακικά τα οποία είναι μόνο παθητικά Έχουμε και μια ομάδα 28 επισκεπτών τους έχει καλέσει ο κύριος Κασίνσκι ο οποίος θα έρθει σε λίγο η επόμενη συνεδρίαση στις 5 Νοεμβρίου δεν θα λάβει χώρα οπότε την επόμενη φορά θα τα πούμε στο Στρασβούργο στις 15 Νοεμβρίου είναι κάτι που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα. Λοιπόν, τώρα για τις διαπραγματεύσεις τις διαθεσμικές έγιναν κάποια πράγματα. Τριμερής διάλογος 8 Οκτωβρίου ε, που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την άδεια πατρότητας ε, μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας από ό,τι φαίνεται όμως το Συμβούλιο είναι αρκετά ακαμπτό στο θέμα αυτό θα γίνει όμως μια νέα συνάντηση στις 6 Νοεμβρίου στον ό,τι αφορά τρίλογο. Τώρα, για τις υπηρεσίες, η ΦΟΠ, ε, η Eurofon, 16 ε, Οκτωβρίου έγινε σχετική συνάντηση. Η Αν Σάντερ θα μας πει δύο λόγια από αυτού. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι, ή είμαι ικανοποιημένη, όπως περιπτώσει εγώ, ε, που υπάρχει συμφωνία στον Τρίλογο, σε αφορά τον κανονισμό για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων ε, σκιωδών εισηγητών, ε, τη γραμματεία ε, της Επιτροπής Απασχόλησης και όλους τους βοηθούς. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά εδώ. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό για όλους, μιας και μας επιτρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου στη λειτουργία του ΣΕΝΤΕΦΟΠ να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια επίσης απέναντι στους συμπολίτε μας. Ένας ε, εμπειρογνώμονας ε, ε, του Κοινοβουλίου θα συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας. Επίσης θα κάνω μια ακρόαση για τον υποψήφιο διευθυντή της υπηρεσίας και βεβαίως κατά την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του οργανισμού θα ακουστεί και η δική μας άποψη. Έχουμε πετύχει πρόοδο και όσο αφορά την των ανδρών και γυναικών ενισχύσαμε και το ρόλο του διευθυντή του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Αυτά για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Τώρα βέβαια θα πρέπει και να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία στην Επιτροπή Απασχόλησης και μετά στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και καλό κουράγιο για τη συνέχεια. Ένα άλλο τρίλογο που ολοκληρώθηκε αφορά το CMD2. Ήμουν εγώ εισηγητή και μπορώ να σας αναφέρω κάποια πράγματα. Φτάσαμε λοιπόν σε συμφωνία με την Αυστριακή Προεδρία. Να θυμίσω ότι είχαμε διακόψει ε, τη συζήτηση του Βουλγαρικής Προεδρίας ε, και το ζήτημα που δημιουργούσε πρόβλημα ε, ήταν οι εκπομπές καπνού ντίζελ έχουμε φτάσει σε ένα συμβασμό ε, που ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις επιθυμίες μας ένα σημαντικό στοιχείο ενδεχομένως το πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, στις παραχωρήσεις που κάναμε αλλά νομίζω πως είναι μια έξυπνη παραχώρηση αυτή για να επιτευχθεί η συμφωνία είναι ότι αφενός θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για το σύνολο του κλάδου δύο έτη για να μπορέσει να προσαρμοστεί και τον τομέα ε, των ε, ε, ορυχείων αλλά και των ε, τούνελ, των εργασιών σε τούνελ, σε σύραγγες, ε, είναι πέντε χρόνια αυτή η μεταβατική περίοδος. Αυτά και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία θα δώσω το λόγο στην κυρία Κινταγιά. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι όπως και όλοι οι υπόλοιποι θέλω ε, να ολοκληρωθεί η νομοθεσία περί προβλέψιμης και διαφανών, και διαφανών συνθήκων εργασίας ε, με μια ευτυχή κατάληξη. Όταν λοιπόν σας, το λέω, σας λέω να αναβληθεί η διαδικασία, αυτό δεν είναι μια απόπειρα να το καθυστερήσουμε εσώ το ολοκληρωθεί η θητεία του Κοινοβουλίου. Και ο ε, Καβέ Σαμπόν έχει κάνει πολλή δουλειά από αυτού του ζητήματο. Όλοι μα το έχουμε κάνει. Όμω ε, νομίζω πω είναι λάθο να ψηφίσουμε επί ενό κειμένου όπου έχουμε 101 σελίδες ε, ο κατάλογος ψήφος, ψηφοφοριών είναι 101 σελίδες και το λάβαμε χθες. Είναι κάπως ηρωνικό να αναμένουμε από, τους, ε, από το προσωπικό μας να δουλεύει όλη νύχτα όταν μιλάμε για μια οδηγία που μιλάει για προβλέψιμες και διαφανείς συνθήκες εργασίας, έτσι. πιστεύω πραγματικά ότι η Επιτροπή απασχόληση ε, πρέπει να δώσει το παράδειγμα του καλού εργοδότη. Έχουμε πλέον μάλιστα σήμερα ε, νέες ε, κοινοποιήσεις, νέες πληροφορίες από τους σοσιαλιστές δημοκράτες που θέλουν ξεχωριστέ ψηφοφορίες. Δεν υπάρχει χρόνος για όλα αυτά. Μπορούμε λοιπόν να το αναβάλουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Γνωρίζω ήμουν και στην Επιτροπή Γεωργίας, ότι συχνά λαμβάνουν χώρα ε, Δευτέρα απόγευμα έκτακτες συναντήσεις, έγινε και την προηγούμενη φορά, ε, όταν ψηφίζουμε επί κάποιων φακέλων ε, που, είναι, που επίγουν για μας. Γιατί δεν κάνουμε και εμείς το ίδιο στην Επιτροπή Απασχόλησης για να εξασφαλίσουμε ότι θα ακολουθεί μια σωστή διαδικασία. Είναι εύκολο να γίνει ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφοριών. Σε μια εκδοχή είχαμε 50 τροπολογίες, μετά είχαμε 117. Ε, δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι σαφή και νομίζω ότι είναι ανεύθυνο να ψηφίσουμε βιαστικά. Οπότε πραγματικά θέλω να σας ζητήσω το θέμα αυτό να το επιλύσουμε συντεταγμένα και λογικά και να ε, αναβάλουμε τη ψηφοφορία για σήμερα. Μάλιστα, υπάρχει αυτό το αίτημα λοιπόν να αναβληθεί η ψηφοφορία. Πρέπει να ψηφίσουμε από αυτού βέβαια. Να πω για τα αιτήματα που υπευλήθησαν ε, για τους συμβαστικούς ε, τους συμβασμούς ε, και τους συμβαστικούς ψηφοφορίες από τους σωστικούς δημοκράτες αποφασίσαμε σε συνεργασία με τη γραμματεία να αφήσουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών ως έχει. Ιδάλλως δεν γίνεται σήμερα. Ε, ξέρω ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις από αυτού σε λίγο. Ε, Επίσης αποφασίσαμε και αρνηθήκαμε ε, τις προφορικές τροπολογίες που προτάθηκαν από το ΕΛΚ. Αλλά θα επανέλθουμε και από αυτού. Τα λέω όλα αυτά για να είμαι σαφής σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία και την ε, αναβολή της ή όχι. Λοιπόν, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε κατά πόσο επιθυμούμε, όπως προτείνει η κυρία επιθυμουμε οπως προτεινει η κυρια μακινιταερ ε, να αναβληθεί η ψηφοφορία. Ψηφίστε ναι λοιπόν αν θέλετε αναβολή. Αν δεν θέλετε αναβολή ψηφίζετε όχι. Άρχεται η ψηφοφορία. That was not clear. Δεν ήταν σαφές ή τουλάχιστον δεν κατάλαβα καλά. Εάν θέλετε ε, να αναβληθεί, ψηφίστε υπέρ. Δεν υπάρχει όμως απάντηση ή αιτιολόγηση στα όσα προτέθηκαν. Ναι, εντάξει, αν κάποιος επιθυμεί να το κάνει. Κύριε Καλβέσαμπον, παρακαλώ. Oui. Χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, ε, ε, ο κύριος Εγώ θέλω απολύτως να σεβαστώ την πρόθεση όλων όσοι θα ήθελαν να αναβληθεί το θέμα. Εγώ θα ήθελα να αναβληθεί για τρεις μήνες γιατί έχω τόσες πολλές ιδέες, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρετε ότι το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. <clears throat> Έχουμε μάθει να δουλεύουμε υποπίεση έτσι κι αλλιώς πρώτον. Δεύτερον, οι τροπολογίες ε, υπάρχουν. Οι συμβιβαστικές έχουν ε, κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, και όλα τα προσχέδια των τροπολογιών έχουν κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν γνωστοποιηθεί και στους σκιώδεις μέσω των πολλών συναντήσεων που είχαμε και χτες το βράδυ απλώς τις χτενίσαμε. και ξέρουμε ότι η γραμματεία όντως δούλεψε ε, με αφοσίωση, ε, δούλεψε ε, τη νύχτα, έστριψε τα μηνύγκια της έτσι ώστε τα πράγματα να προχωρήσουν. Εγώ πάντως έχω εντολή από το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εκπονήσω το, το καλύτερο δυνατό ε, ε, κείμενο. Και όπως είπα και προηγουμένως, το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Και επομένως πιστεύω ότι εντός αυτής της κοινοβουλευτικής εντολής ε, και εντός της θητείας θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εργασία αυτή, γιατί διαφορετικά θα είναι απογοητευτική η εικόνα που θα δώσουμε προς τους Ευρωπαίους εργαζόμενους και μπορεί εδώ να μιλάμε για μια απλή ε, ε, ε, αναπομπή αλλά, αλλά το πονηρό που κρύβεται πίσω από αυτό είναι η αδυναμία να το κάνουμε. Και δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί δεν θα διαβάσω, αλλά και προσπαθώ απλώς να επιχειρηματολογήσω ε, την θέση μου, έστω και αν δεν είναι η θέση την οποία ε, πραγματικά θα ήθελα να πάρω. Γιατί εγώ, αν θέλετε, σε απόλυτο βαθμό θα ήθελα ε, να έχω περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Εγώ είπα από την αρχή στους εσκιώδης ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπροστά μας γιατί έχουμε συγκεκριμένο εγχείρημα να ολοκληρώσουμε και είτε θα μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα κείμενο είτε όχι. Και αν δεν ψηφίσουμε σήμερα θα πρέπει να ψηφίσουμε το Δεκέμβριο. Δηλαδή από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι το Φεβρουάριο θα έχουμε μόνο 6 Φεβρουαρίου για να κάνουμε τον τριμερή διάλογο. Μα αυτό είναι γελίο. Δυστυχώ τα πράγματα δεν είναι ε, ιδεώδη. Πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά εάν θέλουμε να παραδώσουμε κάτι ε, στου εργαζόμενου εντό αυτή τη θητεία πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, Πρόεδρο, ε, μίλησε ένα υπέρ, ένα εναντίον και νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να ψηφίσουμε. Όσοι θέλουν να αναβληθεί η ψηφοφορία θα ψηφίσουν ναι. Όσοι, όσοι, ε, όσοι δεν θέλουν την αναβολή, όσοι δεν θέλουν την αναβολή θα ψηφίσουν όχι. I think, Chair, the, the... Πρόεδρε, νομίζω ότι ε, δεν έχω καταλάβει καλά μέσω της διερμηνίας λέει η κυρία. Εάν θέλετε να ψηφίσουμε σήμερα, θα ψηφίσετε. Αν θέλετε να ψηφίσετε Εάν θέλετε να αναβληθεί η ψηφοφορία θα ψηφίσετε ναι. Πρόεδρος, όσοι θέλουν να αναβληθεί η ψηφοφορία, όσοι δεν θέλουν να γίνει η ψηφοφορία σήμερα, θα ψηφίσουν ναι. Όσοι θέλουν να γίνει η ψηφοφορία σήμερα, θα ψηφίσουν όχι. Καταψηφίζουν την αναβολή. Le vote est Πέρας της ψηφοφορίας, ή μάλλον όχι να ρωτήσω πρώτα, ε, ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 15 ψήφοι υπέρ, 34 κατά, επομένως ψηφίζουμε σήμερα. Alors. Oui, monsieur Rapke. Κύριε Ράπκε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτή δεν είναι... Πρέπει να θέλω να διαμαρτυρηθώ. Ε, έχουμε υποβάλει προφορικές τροπολογίες ε, εντός των προθεσμιών και όμως ε, δεν έγιναν δεκτής. Όσον αφορά αιτήματα των όσον αφορά τις 364, 366, 367 και διάφορες άλλες 798, 051 και 857 πρέπει να σας πω ότι αυτές οι τροπολογίες που όμως έγιναν δεκτές όσο προσθήκες ε, ε, ε, είχαν υποβληθεί εκτός των προθεσμιών και επομένως δεν είναι δυνατόν αυτό να το δεχτούμε διότι αφενός αυτές οι τροπολογίες κατετέθησαν εκτός των προθεσμιών και επίσης αντιτίθενται στο πνεύμα του συμβιβασμού. Είναι απαράδεκτο τέτοιες αλλαγές διαρκής και συνεχής λίγο πριν την ψηφοφορία να εφαρμόζονται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κατανοείτε φυσικά ότι αυτή η ψηφοφορία είναι λίγο περίπλοκη και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ε, κατανοώ αυτά που είπε ο κύριος Ράπκε, αλλά οι τροπολογίες ε, οι οποίες ε, ε, κατετέθησαν αργά από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες δεν έγιναν δεκτές γιατί πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Ξέρω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο αλλά γίνεται δυνατή μια ισορροπία. Δεύτερον, αρνηθήκαμε τις προφορικές τροπολογίες που είχε ζητήσει το ΕΛΚΑ. Είναι σαφές ότι παρά την άρνηση έχουν πάντα την δυνατότητα ε, προφορικά ε, να υποβάλουν την τροπολογία εδώ επί τόπου και αν το κάνετε ε, τότε εγώ απλώς θα πρέπει να επιβεβαιώσω εάν και εφόσον υπάρχουν τρεις βουλευτές που μπορούν προφορικά να τοποθετικούν εναντίον ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες Ανιέσε. Ακούω την αποφασή σας, αλλά πρέπει να απαντήσω στην απάντηση του συναδέλφου. Αυτές ε, δεν ήταν αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες, αλλά τροπολογίες ε, για θέματα που δεν καλύπτονται από τους ε, συμβιβασμούς. Είναι διαφορετικό θέμα το ΕΛΚ έκανε άλλου είδους τροπολογίες. Αλλά οπωσδήποτε ε, εγώ σημειώνω την ε, απόφασή σας. Ναι, δέχομαι την απόφασή σας κύριε ε, Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να ελέγξετε πραγματικά τι συνέβη. Πρέπει να ξέρουμε τι συνέβη. Και επομένως δεν λέω τίποτα μέχρι να μας εξηγήσετε τι θα γίνει με αυτές τις ε, τροπολογίες. Πρόεδρος, η απόφαση ελήφθη. Δεν είναι οπωσδήποτε η πιο καλή απόφαση αλλά σας προτείνω και στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών ε, να μελετήσουμε, να διαρευνήσουμε την κατάσταση και το θέμα αυτό. Πάντως, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία με τον κατάλογο ψηφοφορίας που έχουμε. Εάν κάποια στιγμή υποβληθούν προφορικές τροπολογίες, θα δούμε εκείνη τη στιγμή εάν μπορούν να γίνουν δεκτές ή όχι. Επομένω, στρέφομαι και σε εσά, συνάδελφε, όταν θέλετε να υποβάλλετε κάποια προφορική τροπολογία θα το λέτε και ε, ε, ε, επί τόπου θα δούμε, θα ελέγξουμε αν είναι δεκτή ή όχι. Θα προσπαθήσω να πάω σιγά σιγά. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων γι' αυτό. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν ακόμα στοιχεία τα οποία προσθέθηκαν ε, αργά τη νύχτα ή νωρί το πρωί στον κατάλογο και θα κάνουμε και αρκετέ ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί θέλω τα πράγματα να είναι απολύτω σαφή. Αιτιολογική αναφορά 1, άρχεται η ψηφοφορία πέρας Πέρας. Απερίφθη. Αλλά για κάποιο λόγο δεν το βλέπουμε. Τώρα το βλέπουμε. 5 ψήφοι υπέρ 42 εναντίον. Καμία αποχή. Συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται η συμβιβαστική 29 υπέρ 19 εναντίον. Συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. 39 ψήφοι υπέρ 14 εναντίον. Συμβιβαστική 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπάρχουν ε, ε, πολλές ε, τροπολογίες ταυτόσιμες από την 330 και μετά μέχρι την Γιούρι 43 ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Άρθρο 1, παράγραφος 4, τροπολογία 341 και εδώ έχουμε ε, πολλές ταυτόσιμες τροπολογίες, άρχεται η ψηφοφορία επί όλων αυτών. Πέρας. Απορρίπτονται. Τρία Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 3.49 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Άρθρο 1, παράγραφος 7, αρχική πρόταση κειμένου με, ε, σχετικά με, τον, με το άρθρο και τον κανόνα 174 άρχεται πέρας. Άρθρο 1, παράγραφος 6. Δεν βλέπω σελίδες, λέει ο Πρόεδρος. Αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Για το άρθρο 2, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 51. Συμβιβαστική. Εναλλακτική. Για την ελλογική σκέψη περιθμών 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και έτσι λοιπόν... Να πάμε στο άρθρο 2, παράγραφος 2α ή 411. Βρήκατε παρακαλώ που είμαστε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Ο κ. μου. Να προτείνω το εξή. Να λέτε την ε, σελίδα παρακαλώ, να μας λέτε τη σελίδα γιατί μας βοηθά. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε την ίδια σελίδα. Όχι, όχι, κατάλαβα. Δεν έχετε σελίδε. Όταν ο πρόεδρο λέει τον αριθμό τη σελίδα, θεωρώ γενικά ότι προκαλεί πιο πολλά προβλήματα από τη λύνει. Πάμε στην συμβαστική 11. Και ψηφίζουμε. Περάς. Εγκρίνεται. Γιούρι 53. 54. Έχουμε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα λοιπόν. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Για την 425 ε, έχουμε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 440. Δύο σελίδε παραπέρα. Άρθρο 3, παράγραφο 2, στο σημείο H. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και πάμε παραπέρα. Άρθρο 3, παράγραφος 2, Γιούρι 60. Γιούρι 60. Okay. Le vote est ouvert. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, Οι 485 και 487 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. Τετρακόσια «491» στο σημείο L. «491». Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 493. Άρθρο 3, παράγραφος 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 494 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Στην επόμενη σελίδα. 498. 498-3-2-α. α Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 499. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Η ένα Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Έχουμε τώρα δύο τροπολογίες ταυτόσιμες, η 505 και η Euro 64. Ψηφίζουμε και τις δύο. Πέρας. Απορρίπτεται. 502. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 503. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 504. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 43. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 506. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Can we repeat the votation of... Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία παρακαλώ γιατί δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Ναι, τεχνικό πρόβλημα. Άρα ψηφίζουμε την, ε, την 506 άλλη μια φορά παρακαλώ. 506 ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 508 και 509. Με προφορική τροπολογία της ΑΛΔΕ. Υπάρχουν αντιρρήσεις παρακαλώ για την προφορική τροπολογία. το βλέπω να υπάρχουν ενστάσεις. Άρα ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Europe 65. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάλι έχουμε κάποιες σελίδες να γυρίσουμε και φτάνουμε στο 18. Συμβαστική 18 για το άρθρο 5 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 για το άρθρο 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Ψηφίζουμε. Είναι δύο-τρει σελίδε παραπέρα. Πέρα. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23, άρθρο 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 649. Παραγραφός 2 του άρθρου 8. Ψηφίζουμε. 649. Πέρας. Απορρίπτεται. 29. Με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 9. Συμβαστική 55. Ψηφίζουμε. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρει-τέσσερι σελίδες παρακάτω είναι η συμβαστική τριάτα, παρακαλώ. 24α καινούριο. Συμβαστική 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34 στο άρθρο 11. Ψεφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 36. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 12, 769. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ξαναξεκινήσουμε αμοιάστηκα. Για την 769, παρακαλώ ψηφίζουμε. Le vote est clos. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 7.70 και ΦΕΜ 23 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται ΦΕΜ 22 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται Συμβασμό 37 υπέρ. Ε, άρχιτη ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρα ψηφοφορία Εγκρίνεται. Συμβασμό 38. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. τέσσερι 4-5 ψελίδες πιο κάτω τώρα 813 και η Γιούρι 106. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 814. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 816, 817, 818 και 819 είναι ε, ίδια άρχιτη ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Συμβασμός 39, άρχιτη ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβασμός 40. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Γιούρι 112. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 8.46 Άρχιτη ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας 8.46. Λοιπόν, ξανά άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Και περνάμε τώρα λίγο πιο κάτω. 848 και Γιούρι 114 που είναι τα ίδια. Άρχιτη ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβασμό 41. Άρχιτη ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 859. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 860. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 861. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβασμός 43. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβασμός 44. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 45. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβασμό 46. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβασμό 47. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμό 48. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στα εκτιμώντας. Γιούρι 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται το 1 τώρα άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 77 άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται δύο Τροπολογία 2. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Γιούρι 2. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 80. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. 81. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. ΦΕΜ 3. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορία εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 82. Εκτιμώντας 3. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 83. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 84. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 85. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 86. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Γιούρι 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Γιούρι 3. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Φεμ 4. άρχιτε η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Φεμ 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. ΦΕΜ 6. Ξεχωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Ενενήντα ένα. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 92. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 93. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Γιούρι 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 95. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία Εγκρίνεται. 96. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία Απορρίπτεται. 97. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Γιούρι 5. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 98. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, κυρία Σάντερ, Σάντερ, ναι κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ζητήσω εκ νέου την εισαγωγή μιας προφορικής τροπολογίας για να μπορέσουμε να προσθέσουμε στο συμβασμό, αυτό κάποιες παρεκκλήσεις για τους ε, πυροσβέστες και τους εθελοντές πυροσβέστες. Προφορική τροπολογία λοιπόν. Έχει κανείς αντίρρηση για αυτή την τροπολογία. Ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε δυστυχώ. Συμβασμό 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται. Συμβασμό 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται. Γιούρι 6. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας 6. Τροπολογία 100. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στον συμβασμό 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 117. Εκτιμώντας 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβασμός 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβασμός 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 122 και Γιούρι 9 μαζί, άρχεται ψηφοφορία. Ναι, παρακαλώ. Ένα ερώτημα. Ορισμένε φορέ ψηφίζουμε τροπολογίε οι οποίε είναι παρόμοιε και τι ψηφίζουμε μαζί. Ε, να λέμε ότι είναι ίδιε και διαφορετικέ, το καταλαβαίνω, αλλά που να σχεδόν Πανομοιότυπε δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Είναι σχεδόν πανομοιότυπε, δεν είναι πανομοιότυπε. Ε, κάτι μου διαφεύγει εδώ. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Ναι, από την πρώτη εκδοχή τη ε, του κατάλογου ψήφου λέμε, το λέμε αυτό για κάποιε τροπολογίε γιατί έχουν την, ίδια ακριβώ πρόθεση. Ορισμένε φορέ όμω ε, ε, υπάρχει μια διαφορά σε μία λέξη, χωρί όμω αλλάζει η έννοια. Ε, και σύμφωνα με του νομικού, ορισμένε φορέ ε, κάποια λέξη είναι καλύτερη ε, σε νομοτεχνικό επίπεδο. Ε, όμως η πρόθεση είναι η ίδια ε, και πραγματικά προσέχουμε ιδιαίτερως έτσι ώστε αυτό να γίνει σεβαστό. Δεν υπήρξε δηλαδή καμία αμφισβήτηση από αυτού. Όχι για να σας πειράξει ήθελα απλώς. Έτσι είναι λίγο πειραχτήρι σήμερα ο συνάδελφος. Επόμενη τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Γιούρι 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Le 124, le vote est ouvert. 124 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Θα ψηφίσουμε τώρα το εκτιμώντας 8, δηλαδή τροπολογίες 125 μέχρι και γιούρι 11, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απερίφθησαν. Τροπολογία 130, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 131, υπέρ. Πέρας. Απερίφθη. 132 υπέρ. Πέρας. Ε, δεκτή. 133 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Η 132 εγκρίνεται και περνάμε στην 139. 139, 140, 41, 42, 43. Όχι. Sorry. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, δεν είναι ακριβώς αυτό που είπα. Λοιπόν, να, να ξαναρχίσουμε. Θα ξαναψηφίσουμε την τροπολογία 137. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 137 επί του εκτιμώντας 8. Πέρασε. Απερίφθη. 8 υπέρ. Πέρας. Απερίφθη. 138. Η 138 καταπίπτει 130, 140, 141, 142, 143, 144 και Γιούρι 12 άρχεται η ψηφοφορία επί όλων αυτών των τροπολογιών. Πέρας, δεκτές. 147. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 154. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 10. Υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, γίνεται δεκτή. 157. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 156 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 157 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Γιούρι 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 159. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 12 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 13 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Συμβιβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 17. Είναι δύο σελίδες πιο πέρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 26 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2.35 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 2.36 και Γιούρι 25 από κοινού άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 27 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 28. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Έχουμε μία χωριστή κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα του, της 248 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 248, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Δεκτό το τμήμα αυτό. Τροπολογία που αφορά το τρίτο τμήμα άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 249 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 32. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 33. Άρχεται. Πέρας δεκτή. Συμβιβαστική 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 22. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Γιούρι 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 270. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 266 με προφορική τροπολογία που έχει ζητήσει η Άλντε. Αντιτίθεται κάποιος αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι, άρα την ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 266. Πέρας. Δεκτή. 2.72 άρχεται πέρας απερίφθη Τώρα έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Θα ψηφίσουμε επομένως πρώτα την 273, 274 και Γιούρι 30 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. ΦΑΜ 10 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Δύο ταυτόσημες. 2,75 και 31 γιούρι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Έχουμε τώρα την 276, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 277 είναι προφορική τροπολογία της ΑΛΔΕ. Υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται. Όχι, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή η 277. Περνάμε στην τροπολογία 280. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 280 δεκτή. 281. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 2.84 στην αιτιολογική σκέψη 29 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 285 και Γιούρι 33 ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε λοιπόν από κοινού. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 288 ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. ΦΑΜ 11, ΦΑΜ 11 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 2.89 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 2.91 και 2.92 ταυτόσιμες άρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθησαν χωριστή ψηφοφορία για την Γιούρι 34 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτό το πρώτο τμήμα δεύτερο τμήμα Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. 2.94 και γιούρι 35 ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη σαν. Γιούρι 36. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 42. Άρχεται η ψηφοφορία. περα Δεκτή. 2.98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 2.99 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 300. Άρχεται η ψηφοφορία. δεκτή. 301. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 302. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Γιούρι 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 200, 300, συγγνώμη, 304. Στην αιτιολογική σκέψη 37. Ξαναλέω. Αιτιολογική σκέψη 37 Τροπολογία 304 και Γιούρι 39 ταυτόσημες ψηφίζονται από κοινού, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απερίφθησαν. 305, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 306 άρχεται Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 27. Λέει ο Πρόεδρος, όχι. Τροπολογία 28. Ψηφίζουμε την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Άρα. Στην σελίδα 1 ξεχάσαμε μία τροπολογία είναι η ΦΑΜ 2. Πραγματικά οι δύο πρώτες αράδες. Le vote est ouvert sur le 2. Ψηφίζουμε λοιπόν την ΦΑΜ 2 στην αρχή αρχή του καταλόγου ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Ολοκληρώσαμε λοιπόν. Σας ε, ε, αφήνω ένα-δυο λεπτά στην έτσι ώστε η κάθε ομάδα, αν θέλετε να κάνετε κάποιες ε, διαβουλεύσεις, γιατί ήταν πάρα πολύ περίπλοκη η ψηφοφορία. Όχι, πρώτα όμως να ψηφίσουμε την έκθεση πρώτα. Ψηφίζουμε την έκθεση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, χρειάζεστε λίγο χρόνο, όχι. Όχι, άρα ψηφίζουμε την εντολή. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και γίνεται δεκτή και η εντολή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη ε, για τον χρόνο που ε, μας πήρε αυτή η ψηφοφορία, αλλά ήταν περίπλοκη και έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Thank you, friends, for this... Φίλοι μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ψηφοφορία αυτή και ήταν ε, πολύ δύσκολη, μας ε, ταλαιπώρησε όλους. Να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερής διάταξης, το σημείο 5. Έρασμος. Το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Εμίλιαν Πάβελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το Erasmus Plus είναι ένα από τα πιο επιτυχή ευρωπαϊκά προγράμματα και ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου. Μεγάλη χαρά είναι που είμαι εισηγητής της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό και από ό,τι βλέπετε Είναι φιλόδοξο το σχέδιο γνωματοδότηση που υπέβαλα. Η επόμενη φάση του προγράμματο θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, να επεκταθεί. Όλε οι προηγούμενε άλλωστε εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ζητήσει από την Επιτροπή και τα μέλη να προχωρήσουν πιο δυναμικά το πρόγραμμα αυτό που έχει μεγάλη αντικτύπωση στη ζωή πολλών μα. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, αλλά κυρίως για το μέλλον της Ευρώπης. Πρόκειται για μια επένδυση άλλωστε στην πιο πολύτιμη πρωτεΐλη που έχουμε, τους ανθρώπους μας. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης. Τώρα να τονίσω κάποια θέματα. Καταρχάς το όνομα. Δεν είναι προφανώς ε, μόνο ένα όνομα, είναι και μια ευρωπαϊκή μάρκα, αν θέλετε το Erasmus. Αυτό το Erasmus Plus λοιπόν το υποστηρίζω γιατί περιλαμβάνει όλες τις επιπλέον δράσεις και πρωτοβουλίες του προγράμματος που θα ενταχθούν σε αυτή την ε, περίφημη ομπρέλα. Κατά δεύτερον, υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο που το πω και πιστεύω ότι είναι σημαντικό στοιχείο πέραν από αυτό σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το νέο πρόγραμμα Erasmus Plus θα πρέπει να επικεντρωθεί στην συμπερίληψη και στα άτομα με περιορισμένες ε, δυνατότητες. Επίσης, να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση στο Erasmus Plus, προκειμένου να υπάρξει εκπαίδευση και των πιο ηλικιωμένων σε ό,τι αφορά τα επίπεδα οικονομική υποστήριξη σε ό,τι αφορά επιδοτήσεις, εφαπαξ, ποσά και το καθεξής. Αυτά θα πρέπει να περνούν από τακτική αναθεώρηση και να προσαρμόζονται στο κόστο διαβίωση τη χώρα προορισμού για την ποιότητα, προκειμένου να υπάρχει ο μέγιστος αντικτυπός στους Ευρωπαίους πολίτες θα πρέπει να τονίσουμε την κινητικότητα και την ποιότητα του προγράμματος όπως ορίζεται και στο σχετικό χάρτη κινητικότητας πληροφόρηση, προετοιμασία, αναγνώριση ε, δεξιοτήτων και σαφή προγράμματα εκπαίδευσης. Τέταρτον, επαγγελματική κατάρτιση. Το Erasmus Plus είναι βασικό στοιχείο για τη βελτίωση των ε, καταρτήσεων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται λοιπόν σωστά προγράμματα προκειμένου να υπάρχει α, σωστή αντιμετώπιση. Για διεμάθηση. διαβίου όλοι συμφωνούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα της ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών και θα πρέπει να μπει εγκάρσια σε όλα τα προγράμματα του Erasmus Plus. Έκτον, ίση αμοιβή για την ίδια δουλειά. Αυτή η αρχή θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και στο Erasmus Plus. Ζητάω λοιπόν το προσωπικό όλων των οργανισμών και υπηρεσιών ε, που συμμετέχει στη διαδικασία να έχει την ίδια αμοιβή. Καλώς ορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για πιο πολλές εταιρικές ε, σχέσεις και συνεργασίες για την αριστεία με τα πανεπιστήμια, για παράδειγμα. Πιστεύω όμως ότι μια σωστή γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη είναι βασική απέτηση. Όδων. Και τελευταίο στοιχείο. Αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται από την κινητικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή καταγραφή αυτών και σωστή αναγνώριση τους. Και ζητώ τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη συμμορφώση των συστάσεων του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κατάρτιση και τη μαθητεία, την αναγνώριση των ανεπίσημων και μη δεξιοτήτων, καθώς και όλων των υπόλοιπων ικανότητων που μπορεί να έχει ένα άτομα. Μία τελευταία πρόταση, επιτρέψτε μου. Μου ζήτησε η γραμματεία της ε, Επιτροπής Πολιτισμού να γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Πολιτισμού του Δεκέμβριου. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις ε, συζητήσεις και τις συμβαστικές προτάσεις που θα καταφέρουμε να βρούμε μετά την προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Αν κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας, νομίζω τα θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο και όχι τον Φεβρουάριο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα το κρίνουμε όταν ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολή των τροπολογιών την Τρίτη. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία και μαζί σα και με όλους τους σκιώδει για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι αν πετύχουμε ποιοτική εφαρμογή του Erasmus Plus θα έχει μεγάλη και θετικό αντικτύπο σε όλους μας τους πολίτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πάβαλη. Το λόγο έχει ο κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο τον κύριο Πάβελ ε, για την επεξεργασία του θέματος και για την ε, παρουσίαση. Νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι εφικτό. Σε ό,τι αφορά την ενισχυμένη συνεργασία σε όλες τις ε, σε όλα τα τμήματα αλλά σε κάθε περίπτωση να υπάρχει και σωστή εκπροσώπηση της Επιτροπής μας. Χθε έγινε μια ακρόαση της Επιτροπής Πολιτισμού, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και διαπιστώνουμε πόσες ιδέες είναι ταυτόσιμες. Θα θέσουμε προφανώς και έμφαση σε διάφορα σημεία για το Erasmus Plus. Σίγουρα είναι ένα από τα ορόσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το συν λοιπόν αυτό το πλάσ αυτό θέλουμε να δείξουμε πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε τους νέους. Όχι με κενά λόγια, αλλά με συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Η κινητικότητα είναι όλο και πιο σημαντική και όταν υπάρχουν εμπόδια θα πρέπει να προσπαθούμε να δίνουμε τις σωστές απαντήσεις. Ενίσχυση λοιπόν των αρμοδιοτήτων, συμφωνούμε. Θέλουμε να τονώσουμε την απασχολησιμότητα των νέων. Αυτό φυσικά το βοηθάει ιδιαίτερα το Εράσμος και αυτή η έλλειψη μέλλοντος που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι. Θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται με προγράμματα όπως αυτά του Erasmus Plus. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι. Εγώ χαίρομαι που ο κύριος Ότινγκερ, ο Επίτροπος για τα θέματα προπολογισμού, είπε ότι με όλες τις περικοπές που γίνονται να μην γίνει περικοπή σε ένα θέμα μόνο, το Erasmus Εδώ θέλετε διπλασιασμό των πόρων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε σίγουρα την τάση αυτή. Τι μπορεί να πετύχει λοιπόν το Erasmus σε αυτή την εποχή της ε, ανεργίας των νέων, τι θα πρέπει να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε. Το Erasmus Plus θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα πρόγραμμα υποστήριξη των φοιτητών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερο κύρος για την επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλάβουν οι νέοι στα πανεπιστήμια και σε όλε τι σχολέ ότι το Erasmus Plus απευθύνεται σε αυτού. Και επίση οι πόροι του Erasmus θα πρέπει να δαπανηθούν για την καταπολέμηση του λαϊκισμού, προκειμένου να προωθήσουμε πιο πολλά δημοκρατικά έργα για να καταλάβουμε τι ακριβώ είναι το επικίνδυνο στη ριζοσπαστικοποίηση, στο λαϊκισμό, στην περιθωριοποίηση, για να αποκτήσουμε ακριβώ λοιπόν μια τέτοια συνειδητοποίηση, μια τέτοια αντίληψη, μια τέτοια νοοτροπία θα πρέπει να τονίσουμε το Erasmus Plus, γιατί πρόκειται για ένα γενικότερο πρόγραμμα κατάρτιση και εκπαίδευση και γενικότερη παιδεία. Τα προγράμματα συμπερίληψη, σύμφωνα μαζί σου, Εμιλιάν, θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε και θα πρέπει να κρατήσουμε και τον κόκκινο μύτο, αν θέλετε, το, το, το στοιχείο αυτό που ενώνει όλες τις δράσεις. Σίγουρα θα καταθέσω κάποιες σχετικές τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά νομίζω ότι η έκθεση θα είναι καλή και βάσει και αυτών που μας είπε συνάδελφε, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε σε μεγάλο βαθμό και έτσι ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε με μία φωνή, κυρίως για να μην έχει την εντύπωση ο οποιοδήποτε νέος ότι τον αφήνουμε στην τύχη του, μόνο του. Όχι. Να τους δείξουμε στους νέους ότι θέλουμε να αναπτύξουμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα προσόντα τους. Και εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε οικονομικά προς την κατεύθυνση αυτή και εγώ προσβλέπω στη συνεργασία μας, λοιπόν. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η άλλη εκπροσωπείται από την κυρία Στίβενς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πολύ καλή δουλειά. Και είμαι πεπισμένη ότι θα αποτελέσει αυτό μια σωστή βάση την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε σε μια ισόρροπη και θετική συμβαστική λύση. Το πρόγραμμα Εράσμους είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό. Δίνει στον κόσμο μοναδικές ευκαιρίες για να αποκτήσει πραγματικά δεξιότητες και ικανότητες που θα δώσουν τελικά προβάτισμα στην αγορά εργασίας. Όποιος έχει περάσει από τη διαδικασία Εράσμους βρίσκει πιο εύκολα δουλειά. Τα στοιχεία μιλούν από μόνος τους. Ε, οι επενδύσεις στην παιδεία είναι επενδύσεις που ε, έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Προτείνω λοιπόν ε, σημαντική αύξηση του, της χρηματοδότησης ε, του Εράσμους, γιατί χρειαζόμαστε επιπλέον κονδύλια. Είναι μεγάλη ζήτηση. Θα πρέπει να γίνει εσωτερική ανακατάταξη της χρηματοδότησης, πιστεύω. Και χαίρομαι που ο συγητής ε, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ε, προσβασιμότητα του προγράμματος Εράσμους για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί εδώ υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ακόμα. Ένα παράδειγμα το οποίο γνωρίζω εγώ από την ίδια εμπειρία μου είναι η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση που υπόκειται η κοφή για να επικοινωνούν μέσω νοηματικής. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και να πω ότι το πρόγραμμα το πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ε, προδιαγραφές του χάρτη του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Και επίσης ε, με απασχολεί το θέμα των ε, επαγγελματικών δεξιοτήτων. Θα πρέπει να γίνονται λοιπόν θετικές επιλογές. Θα πρέπει να δίδεται η σωστή εκπαίδευση για κάθε μαθητή και, και φοιτητή προκειμένου να έχει τη σωστή ανάπτυξη Επίση, εκτιμώ το γεγονό ότι ο εισηγητή επιμένει στο θέμα τη ποιότητα. Γιατί στο παρελθόν θεωρώ ότι είχαμε εστιαστεί υπερβολικά σε ποσοτικού στόχου. Το θέμα δεν είναι μόνο πώ οι φοιτητέ συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εράσμου. Και η πρωτοβουλία Discover EU. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν είναι ο Άι Να εκφράσω μερικές ανησυχίες μου. Δεν είμαι υπέρ της συγκεκριμένης ανάθεσης χρηματοδοτήσεις και κονδυλίων σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους ετούντες άσυλο, θεωρώ ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να υπάρξει ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών και να ε, υπάρχει διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Αυτό είναι το πιο λογικό θεωρώ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι η εκπαίδευση αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήμουν πιο προσεκτική με την ιδέα της Ευρωπαϊκής, ε, των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είμαι υπέρ μια πιο ε, εντατική συνεργασία μετα, μεταξύ των πανεπιστημίων. Προσβλέπω στην μελλοντική επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και με τους κοιότητες εισηγητές και νομίζω ότι τελικά η γνωμοτότηση αυτή θα είναι περίφημη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Stevens. Ευχαριστώ την κυρία Stevens. Και τώρα η κυρία Λαμπάντιοβα δεν είναι εδώ όμως. Είναι κάποιος άλλος εδώ που να εκπροσωπεί την Άλντε. Όχι, να περάσουμε στην Κούε τότε. Ο κύριος Λεγιαρίκ δεν είναι εδώ. Κάποιος άλλος από την Κούε τον αντικαθιστά. Όχι. Πάμε στους πράσινους λοιπόν. Ο κύριος Μέσεριτς και αυτός λείπει. Πάμε λοιπόν τώρα στην ENF. Η κυρία Μελά είναι εδώ, ούτε αυτή. Μάλιστα. Ίσως ο κύριος Πάβελα θέλει να προσθέσει κάτι για να κλείσουμε με το θέμα. Στα γερμανικά να επιχειρήσω. Ε, επειδή ήταν και μεγάλη ψηφοφορία, προφανώς οι συνάδελφοι ε, έπρεπε να φύγουν και δυστυχώς δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θα τα δούμε και με τους κοιόδης. Προκειμένου το Erasmus Plus να μπει στην προπτική που του αρμόζει. Να είναι θετική η παρουσίασή του και η διαμόρφωσή του και περαιτέρω να διορθωθεί. Δύο-τρία στοιχεία να πω σε σχέση με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Τριπλασιασμό προφανώ είναι δύσκολο. Τριπλασιασμό των κονδυλίων. Αλλά το Κοινοβούλιο πιστεύω στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει με μια εντολή, με την εντολή που του δώσαμε για τον διπλασιασμό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ξεκινήσουμε ζητώντα τριπλασιασμό, είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα πετύχουμε το διπλασιασμό που επιθυμούμε τελικά. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά το λαϊκισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση που μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε με το Erasmus+. Plus. Κάτι που μπορούμε να βελτιώσουμε είναι τον πολυσύνθετο χαρακτήρα. Γιατί αυτό πολλούς αποτρέπει να κινηθούν προς την ε, πλευρά του Erasmus γιατί υπάρχει μεγάλο γραφειοκρατικό άγχος. Η κυρία Στίβενς έθεσε το θέμα της ποιότητας ε, και το αντιπαρέθεσε με την ε, ποσότητα. Εδώ να πούμε το εξής. Όταν επιθυμούμε τριπλασιασμό των φοιτητών που ωφελούνται των δικαιούχων δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με διπλασιασμό των κονδυλίων. Σε ό,τι αφορά το Discovery U, δεν το επέκρινα ως πρόγραμμα. Είπα απλά ότι θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο το καλωσορίζω, να φροντίσουμε να περιλαμβάνει και ένα πολιτισμικό σκέλος, προκειμένου αυτοί που χρησιμοποιούν πόρους του να μην επιστρέφουν στα σπίτια του μόνο με μια ωραία φωτογραφία. Να ζήσουν πραγματικά τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός μας ενώνει και αυτό θα πρέπει να το μεταφέρουν στις πατρίδες τους και να το διαβιβάζουν και περαιτέρω σε όλους τους υπόλοιπους γνωστούς τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και προσβλέπω στη συνεργασία μας και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να ψηφίσουμε τον Δεκέμβριο. Thank you. Deadline for amendments. Ευχαριστώ. 23 Οκτωβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες το μεσημέρι και ψηφοφορία στις 22 Ιανουαρίου ε, στην Επιτροπή μας και τον Φλεβάρι ε, στην Επιτροπή Κούλτ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 6 της μέσης διάταξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, ESF Plus. Είναι στην ημέρα στη διάταξη όλων των πολιτικών ομάδων το θέμα αυτό. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Λόπεθ Φοντανιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι στην Επιτροπή μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόθεση της απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη. Ως μέλη της Επιτροπής αυτής, καθήκον μας είναι να συνεχίσει να παίζει αυτό το ρόλο και για την περίοδο 2021 έως το 2027. Η σημασία της ε, έκθεσης αυτής ε, έχει αποδειχθεί και από τις 768 τροπολογίες που υπευλήθησαν. Είμαι βέβαιο ότι θα συνεισφέρουν στην βελτίωση του προτινόμενου κειμένου όπως ήδη έχουμε πει, έχουμε λίγο χρόνο για την έγκριση της έκθεσης. Θα την ψηφίσουμε στις 26-27 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια ε, αποσαφήνισης στις διαπραγματεύσεις για να διαδικηθούμε σε ένα κείμενο το οποίο είναι χρήσιμο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Για την ώρα είχαμε δύο συναντήσεις των σχεδόν εισαγητών, Προέπεται και μία συνάντηση κάθε εβδομάδα έως τις ψηφοφορίες. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ καλό το κλίμα στις συναντήσεις αυτές, κάτι που αποδεικνύει ε, ότι υπάρχει βούληση να φτάσουμε σε συμφωνία. Το πιο περίπλοκο σημείο, αυτό που δεν έχουμε ακόμα αγγίξει κιόλα, είναι το, η αναφορά στο άρθρο 7 ε, για την θεματική συγκέντρωση. Ε, όπως έκανε και κατά την παρουσίαση της έκθεσης πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τη διασύνδεση μεταξύ των ε, συστάσεων αναχώρα και του Ευρωπαϊκού, Κοινωνικού Ταμείου Plus. Ε, είναι αναγκαίο αυτό για ε, να μπορέσει να προχωρήσει ο κοινωνικός πυλώνας και μέσω των συστάσεων αναχώρα αν μπορούμε να εντοπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα και αυτό θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τις αρχές που διέπουν τον κοινωνικό πυλώνα. Ο κοινωνικός πυλώνας είναι αυτός ο οποίος θα, ε, θα εφαρμόσει την πραγματικότητα τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα κράτη-μέλη από εκεί και πέρα πρέπει να έχουν μια ευελιξία για να μπορέσουν να διαθέσουν τους πόρους στους τομείς εκείνους όπου είναι αυτό περισσότερο αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, ε, τις τοπικές, τις περιφερειακές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτό είναι άλλο ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να υποτελέσει αντικείμενο συζήτηση στις ε, συζητήσεις μας, στις επαφές μας. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ορίζουμε ποσοστά για διάφορους θεματικούς τομείς, ε, θεματικές ενότητες. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει ένα σημαντικό ποσοστό για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη. Χθες, 17 ε, Οκτωβρίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την εκρίζωση της φτώχειας. Η φτώχεια είναι ε, ένα κακό το οποίο καταστρέφει την κοινωνική συνοχή. Επίσης, 85% ε, πρέπει να είναι χρηματοδότηση για να επιτευχθεί ο στόχος ε, ε, υπαριθμών 11, να καλυφθούν ε, δηλαδή βασικές ανάγκες και να συνοδεύεται αυτό ε, για με από πολιτικές για την ένταξη των πλέον μειονεκτούσων ομάδων. Ταυτόχρονα συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να παραμείνει η απασχόληση των νέων ως βασική προτεραιότητα των Ευρωπαίων. Ταυτόχρονα πρέπει να βρεθεί μια σημεία ισορροπία όμως, διότι αν προκαθορίσουμε κάποια ποσοστά πολύ υψηλά, υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουμε χωρίς χρήματα για άλλες ε, δραστηριότητες και άλλα μέτρα τα οποία είναι και αυτά απαραίτητα. Είμαστε λοιπόν στο σωστό δρόμο πιστεύω. Αν συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ε, όπως ε, έχει γίνει, ε, έχει λάβει χώρα αυτή ως τώρα, πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα τύχει της υποστήριξης της ευρείας πλειοψηφίας των μελών μας, κάτι το οποίο ελπίζω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Έρχεται όπου να είναι. Είδα τον βοηθό του. Θα τον περιμένουμε λοιπόν. Και εντωμεταξύ θα το λόγο στην κυρία Τρεμπέσιους, την οποία όμως ε, ε, αντιπροσωπεύει η κυρία Μακιντάιερ. Παρακαλώ κυρία Μακιντάιερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω βεβαίως ε, εξ ονόματος του, του, της εσκιώδους ε, εισηγήτριας που δυστυχώς ε, δεν είναι εδώ, αλλά μου άφησε κάποιες σημειώσεις. Μου λέει λοιπόν ότι αρχικά το προσχέδιο του κειμένου φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με ιδέες οι οποίες υποστηρίζονται από την πολιτική μας ομάδα. Θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινωνικό Ταμείο Plus ε, μπορεί να αποτελέσει όχημα καλύτερης αποτελεσματικότητας ε, και ε, δικαιότερης κατανομής πόρων εκεί που περισσότερο χρειάζονται και που μπορούν να δώσουν περισσότερη προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, στη συζήτηση για τις συμβαστικέ τροπολογίες φαίνεται να προκύπτουν αρκετά ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Ε, οι συμβαστικές τροπολογίες ε, πρέπει να οδηγούν ε, σε ε, μεγαλύτερη περιπλοκότητα που αντιτίθεται στην αρχική ιδέα της απλούστευσης. Επίσης, ε, όταν τα κράτη-μέλη μπορούν να κατανείμουν τα κονδύλια ε, ανάμεσα σε διάφορες πολιτικές, αυτό όντως αποτελεί πολύ μεγάλο στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν υπό την αρχή της μοιρασμένης διαχείρισης τα κράτη-μέλη να έχουν την δυνατότητα, την ευχέρεια να αποφασίζουν. Πιστεύουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ε, δώσουν περισσότερη χρηματοδότηση ε, σε παιδεία τα οποία θεωρούν ε, πλέον απαραίτητα. Επίσης, να μην λησμονούμε ότι υπάρχουν ταμεία όπως ας πούμε το Ταμείο για τους Φτωχότερους που ε, έχουν στόχο την καταπολέμηση της ένδυας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν ε, το ε, ΕΚΤΑΦ θα πρέπει να αφορά περισσότερο συγκεκριμένες δράσεις ναι, για την ανεργία, την απασχόληση, την εκπαίδευση αλλά ε, και την ε, διοικητική ε, διαχείριση και όχι μονάχα να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης δεν είναι δυνατόν κανδύλια από αυτό το ταμείο να πηγαίνουν προς την παράτυπη μετανάστευση γιατί υπάρχουν άλλα ταμεία τα οποία χρηματοδοτούν ακριβώς αυτό το στοιχείο της μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Μακεντάιαρ. Είστε έτοιμος κύριε Μποναφέη. Έχετε το λόγο λοιπόν αφού είστε έτοιμος. Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Είχα την εντύπωση ότι δεν είχαμε φτάσει ακόμα στην εξέταση αυτού του σημείου. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο λοιπόν στις 768 τροπολογίες ε, που έχουν υποβληθεί όσον αφορά το ACT ε, μπορούν να βρεθούν ε, πολλά σωστά εναλλακτικά στοιχεία σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια που με τρόπο ταχύ και οργανωμένο προχώρησε στη συζήτηση των συμβαστικών τροπολογιών δείχνοντας μέχρι τώρα μεγάλη διάθεση εξέβρεσης ε, ε, ευρείας πλειοψηφίας. Ε, είναι σημαντικό να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι με ευρεία εντολή έτσι ώστε και το παρόν κοινοβούλιο αλλά και ε, οι δικαιούχοι, το, οι τωρινοί και οι μελλοντικοί πραγματικά να έχουν να αντιμετωπίσουν μια Ευρώπη η οποία θα είναι καλύτερη, θα είναι ένας καλύτερος τόπος ζωής ε, ε, που θα έχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποια πιο περίπλοκα στοιχεία τα οποία θα συζητηθούν την άλλη εβδομάδα, ας πούμε άρθρο 7 όσον αφορά την θεματική συγκέντρωση, 9 για τη φτώχεια, 10 για την ε, υποστήριξη της ε, ε, νεανικής απασχόλησης, καθώς επίσης και άρθρο 11 συστάσεις αναχώρα εντός του εξαμήνου του Ευρωπαϊκού Εξιαμήνου. Οι τροπολογίε που υποβάλλουμε ω σοσιαλιστέ και δημοκράτες ε, ε, προσπαθούν να κάνουν πιο ευρύ το πεδίο, προσπαθούν να αυξήσουν το ποσοστό τουλάχιστον στο 30% όσον αφορά του εθνικούς ε, πόρους και βεβαίως χρηματοδότηση της καταπολέμησης ε, των ε, υλικών στερήσεων. Επίσης, όσον αφορά την υποχρέωση δαπανών των κρατών μελών για την νεανική ανεργία. Υπάρχει βέβαια και μία σχετική πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που ε, θέτει ως πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς αυτή την καταπολέμηση της, ευρωπαϊκής, της ε, ανεργίας των νέων. Υπάρχει όμως και η υλοποίηση της, ε, του προγράμματος για τους νέους που είναι η εγγύηση για τους νέους. Επίσης, αν θέλουμε να βελτιώσουμε πραγματικά την μακροοικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, το πρόβλημα ε, βλέπουμε ότι δεν λύνεται όσον αφορά αυτό το μεγάλο πρόβλημα της νεανικής ανεργίας. Η ανεργία των νέων είναι θέμα ιδιαίτερος προσφυλές. Ε, στην ομάδα μου μας προβληματίζει πολύ και πιστεύουμε ότι θα πρέπει εντός του κοινωνικού ταμείου ε, θα πρέπει να βρει μια θέση αντίστοιχη αν όχι μεγαλύτερη από αυτήν που είχε στο προηγούμενο ταμείο έτσι ώστε να μπορέσουμε και μέσω συνεργειών να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το Child Guarantee τώρα, εγγύηση για τα παιδιά. Πρόκειται για μια δομή που προτείνεται από την Επιτροπή στην, ε, ε, προβλέποντας συγκεκριμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένη αναφορά εντός του άρθρου 1. Συζητήσαμε πολλές φορές το θέμα αυτό μέσα από πολύ ζωντανέ συζητήσεις. Δουλέψαμε εντελεχώς με υπηρεσίες και οργανισμούς και οργανώσεις που υποστηρίζουν τα παιδιά. Θεωρούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από τη δική μας Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ε, στους ε, πολίτες μας ε, με το πέρας αυτής της θητείας. Ένα μήνυμα ισχυρό υπέρ των παιδιών και για την προστασία των παιδιών. Κάνω έκκληση λοιπόν στους συναδέλφους και στην εισηγήτρια να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε πιο καλές λύσεις γιατί γνωρίζουμε ότι η πρόταση μπορεί να γίνει μέσα από την πολύτιμη συμβολή όλων. Μπορεί να γίνει, λέω, μια εξαιρετική πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπονιφάη. Η κυρία Σελίμοβιτς, από την Άλντε, παρακαλώ. Ο κύριος Σελίμοβιτς, ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία της, ε, ε, την οποία είδαμε και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις των σκιωδών. Θα κάνω κάποιες, ε, κάποια γενικά σχόλια και μετά θα πω και κάποια πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω την ανάγκη κοινωνικής ένταξης ε, όσον αφορά τους μετανάστες στο ΕΚΤ Ξέρω ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις σχετικά με τους πρόσφυγες και την προσφυγική κρίση. Ξέρω ότι ε, ξεκινάμε από διαφορετικά σημεία, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι είτε σας αρέσουν ή όχι οι πρόσφυγες, είτε είστε υπέρ ή όχι, θε, τους θέλετε εδώ ή τους θέλετε μακριά, είτε θέλετε ανοιχτά ή κλειστά σύνορα, ή δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη εδώ και δεν είναι δυνατόν ε, να μην βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ενταχθούν στην κοινωνία. Όποια και αν ήταν η θέση του καθενός στη διάρκεια αυτής της προσφυγικής κρίσης, τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ και επομένως θα πρέπει να τους εντάξουμε στις κοινωνίες μας. Κατά την έννοια αυτή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη μέτρων κοινωνικής ένταξης. Δεύτερο, Υποστηρίζω ιδιαίτερα την ιδέα ε, των κρατών που θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την νεανική ανεργία. Είχαμε προβλήματα με την ανεργία των νέων και πριν από την ε, κρίση. Είναι ένα πρόβλημα που σοβεί στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. και τώρα τα, οι αριθμοί έχουν αυξηθεί λόγω της κρίσης. Επομένως θα πρέπει να υποχρεώσουμε, να πιέσουμε μάλλον τις χώρες να κάνουν ε, περισσότερο για αυτήν την ε, ομάδα ε, των νέων που δεν έχουν ούτε δουλειά ούτε βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση. Τα, η, ομάδα NET όπως λέμε πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν ο καθένας να προσπαθεί να μπλοκάρει ας πούμε ε, κάποιους πόρους. Ε, μπορώ να σεβαστώ την ιδέα ότι καθένας θέλει να προστατέψει κάποιες ε, τάξεις ή κάποιες ομάδες αλλά πραγματικά στο τέλος ε, θα φτάσουμε σε καταστάσεις τις οποίες δεν θα μπορούμε να προβλέψουμε. Δεν θα είναι οι πρόσφυγες, δεν θα είναι η Ελλάδα, δεν θα είναι ε, η συγκεκριμένη κατηγορία, θα είναι κάτι άλλο. Ε, καταλαβαίνω ότι ο καθένας είναι, είναι κάπως λογικό να προσπαθεί ο καθένας να κρατήσει για τον εαυτό του τους πόρους αλλά και τα κονδύλια, αλλά πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω τους συναδέλφους να δείξουν κάποια ευελιξία τουλάχιστον για ορισμένα τμήματα των, της χρηματοδότησης συγκεκριμένα θέματα. Ε, το ε, διοικητικό άκθος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μείνει όσο γίνεται πιο χαμηλό. είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το βάρος το διοικητικό είναι απίστευτα βαρύ. Δεύτερο, ε, διακριτική μεταχείριση. Το έχω ξαναπεί και σε άλλες συνεδριάσεις. Ε, κάποιες χώρες έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ε, στην Σουηδία είμαστε πολύ ξεκάθαροι όσον αφορά τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις. Αλλά εάν μιλάμε για συγκεκριμένα στοιχεία επί τη βάση των οποίων γίνεται διακριτική μεταχείριση, τότε... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούμε και το λέω για τους Σουηδούς από όλε τις ομάδες. Ε, φαντάζομαι ότι και οι άλλες χώρες έχουν περίπου ίδια προβλήματα, δηλαδή θα πρέπει η διατύπωση να είναι τέτοια, ώστε να βρούμε λύσεις που να είναι αποδεκτές από όλους. Έχω και κάποια άλλα θέματα να αναφέρω. Κανένα πρόβλημα η σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλά να μην λησμονούμε ότι η συμβολή ε, αυτού του ταμείου είναι να λύσει κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει ε, να ε, απολυ... θα πρέπει σε απόλυτους βαθμούς αυτές, αυτά τα θέματα να τεθούν ως προτεραιότητα. 15% του ε, Ταμείου ε, στο Shared Management για την αντιμετώπιση της ε, νεανικής ανεργίας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν θέλω, καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει ο καθένας να κρεμάσει σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το κείμενο οτιδήποτε επιθυμεί και να το κάνουμε τελικά χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να περιλαμβάνονται και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Εγώ σας ευχαριστώ. Η Γαμπριέλ δεν είναι εδώ, αλλά την ε, αντικαθιστά η κυρία Όιλαντ. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω ε, συγγνώμη εκ μέρους της Γκάμπι Τζίμερ που δεν είναι ε, εδώ και θα παρουσιάσει το θέμα εξ της στην ΓΚΟΕ. Ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ε, Ταμείου γιατί πραγματικά μπορεί να σημάνει πολλά για τους πολίτες σε ε, ολόκληρη την Ευρώπη. Θα μπορεί να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν οικονομικά και άλλα προβλήματα κυρίως αν αναφερόμαστε στους πιο στερημένους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αρκετές τροπολογίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα ας πούμε να φτάσει το όριο για την φτώχεια στο 30% ε, ε, το, το, το, το, κομμάτι που θα πηγαίνει στην καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι, τα παρόντα στοιχεία για την κοινωνική συμπερίληψη και να μείνουν τουλάχιστον στα όρια του προηγούμενου. Δεν θέλουμε καμία ε, αναφορά ε, με το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο οι συστάσεις του εξαμήνου θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορούν συγκεκριμένους μακροοικονομικούς στόχους και επομένως ενδεχομένως δεν θα βοηθήσουν τους πιο στερημένους και αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης είναι υπερβολικά κεντρικές όλες οι προτάσεις αυτές και επομένως δεν αφορούν πραγματικά πραγματικά ενωσιακή προσέγγιση. Επίσης η συνάντηση ας πούμε μεταξύ κυβερνήσεων, εκπροσώπους εργαζομένων Κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να είναι ε, πραγματικά σωστή και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κώδικας δεοντολογίας καθώς επίσης και ε, το κεφάλαιο 6 του κοινού προγράμματος. Ε, πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει το σύστημα reporting να παραμείνει όσο γίνεται πιο απλό και επομένως να μην υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση. Επίσης για το παράρτημα 2 έχουμε υποβάλει τροπολογία έτσι ώστε ε, να ε, μην υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να αποκαλύψει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης θεωρούμε ότι ε, μπορούμε να κάνουμε μια νέα προσέγγιση με βάση νέων προτάσεων. Καλή τύχη λοιπόν και στην εισηγήτρια ε, και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει και η συνεργασία έτσι ώστε το κείμενο το τελικό να είναι καλύτερο από το αρχικό. Ευχαριστώ πολύ. The Greens, Thank you, Η πράσινη. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι αναφέραν πολλά στοιχεία. Θα είμαστε σύντομοι. Πέντε βασικούς στόχους έχουμε, τους οποίους θα θέλουμε να θέσουμε στη συζήτηση σε ό,τι αφορά και τους πόρους για την κοινωνική περίληψη στο ΕΚΤΕ δεν είναι μόνο ένα ταμείο με το οποίο μοιράζουμε χρήματα. Όχι, θέλουμε να πετύχουμε και κάποιους στόχους και πιστεύω ότι η κοινωνική περίληψη συμπερίληψη είναι ένας από τους βασικούς στόχους και πιεστικούς, τα πιεστικά προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δεύτερο επίπεδο, οι περιθροποιημένες ε, κοινότητες Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες χρήζουν ε, πιο ειδική προσοχή και στην Επιτροπή Ρέτζη κάναμε μια σχετική ακρόαση και το ESF, το ΕΚΤ, ήταν ένα πρόγραμμα στα οποία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 2% θα πρέπει να αναφέρεται σε περιθωριοποιημένες ε, ομάδες. Επόμενο θέμα, το θέμα της προσέγγισης των θεμελιδών δικαιωμάτων. Θα θέλαμε το ΕΚΤ να χρησιμοποιείται μόνο για προγράμματα τα οποία δεν είναι ενάντια με τον χάρτη ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάναμε κάποιες παρατηρήσεις ότι στο παρελθόν είχαμε χρηματοδοτήσει δράσεις οι οποίες είναι κατά ουσιαστικά της υλοποίησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να μην συμβεί αυτό στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Τέταρτο σημείο. Η σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σε ό,τι αφορά και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι το ΕΚΤΕ Plus ε, μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου ο πυλώνα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων να είναι πιο απτό, πιο προσιτό για τον πολίτη. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτού του πόρου για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Και τελευταίο σημείο από πλευρά δική μου, μια και είμαι από μια περιφέρεια που αντιμετωπίζουμε μεγάλε προκλήσει ε, μεταβατική φύση, θα έλεγα να θέσουμε το ζήτημα της α, δίκαιης μετατροπής μιας περιοχής, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που μας απασχολούν, θέματα απασχολησιμότητας, δεξιοτήτων και πολλά άλλα τέτοια δίκαια αιτήματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσει αυτή τη δίκαιη μεταμόρφωση των περιοχών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Αγγία δεν είναι εδώ. Από το EFTD. Δεν την αντικαθιστά και κανένας από ό,τι βλέπω. Ούτε η κυρία Μπιζότο από το ENF είναι εδώ. Και άρα περνάμε στα μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Περίνσκι, καταρχάς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. σε ό,τι αφορά την ε, περίοδο μετά το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την απλοποίηση. Κατανοούμε ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό ε, των διαφόρων εργαλείων προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο δεν ε, κατάφερε να προτείνει και να συμπεριλάβει διατάξεις στο μελλοντικό κανονισμό του ΕΚΤ που θα δημιουργήσουν ένα σαφές πλαίσιο και που θα εξηγήσουν καλύτερα πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν ως τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε για να πετύχουμε τις πολιτικές αυτές, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά τη συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρόλος λοιπόν του ταμείου αυτού, του Ταμείου Κοινωνικής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Γι' αυτό λοιπόν βασιζόμαστε σε πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα στοιχεία αυτά λοιπόν ελπίζουμε ότι θα είναι πιο κατανοητά από τον πολίτη και θα ανταποκρίνονται πιο πολύ σε αυτά που αναφέρονται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άλλα δύο στοιχεία τα οποία αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το Κοινωνικό Ταμείο και το θέμα της υγείας. Αυτά θα συμβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Συνοχή, αλλά δεδομένη τη ελάχιστη χρηματοδότηση δεν ξέρουμε τι ακριβώ θα πετύχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να οριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια τη κοινωνική συνοχή με καλύτερο τρόπο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μια μικρή παρένθεση Επιτρέψτε μου για να αναφέρω το εξή. Οι συστάσει σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θεωρώ ότι αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τι ε, προτεραιότητε τη κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε μια επιφυλακτική στάση σε ό,τι αφορά τι συστάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. για να μην στραφούμε προς μία κατεύθυνση την οποία δεν επιθυμούμε σε ό,τι αφορά την ε, αντικατάσταση της πολιτικής συνοχής από μία οικονομική πολιτική εμ, ε, συντονισμού. Κάθε χρηματοδότηση έχει το στόχο της, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να θέσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τους στόχους σε ό,τι αφορά τα τρία στοιχεία της ε, Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Υπάρχουν ουσιαστικά οι δραστηριότητες. όπως το παρελθόν, αλλά δεν θα καλυφθούν νέες ε, ανάγκες. Και δεν υπάρχει συντονισμός με την τρόπο. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που έχουμε πετύχει τώρα. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν ε, επακριβείς στόχοι, ε, επιχειρούμε να επιστήσουμε την ε, προσοχή λοιπόν όλων προς το κενό αυτό και ελπίζουμε μετά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να έχουν καλυφθεί αυτά τα κενά. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αντί να προτείνουμε κονδύλια για κάθε στόχο, προτείνεται μεταφορά πόρων από άλλες ε, πρωτοβουλίες. Και κατευθυνόμαστε προς την ε, ε, άμεση διαχείριση. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό ταμείο περιλαμβάνει πολύ χρήσιμα στοιχεία τα οποία σίγουρα θα αξιοποιηθούν για λειτουργικέ δράσεις και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κανονισμό για το Ταμείο να είναι υποκίνητη διαχείριση και να ορίζει με σαφήνεια τους κανόνες Το έγγραφο απευθύνεται και σε κάποιες τεχνικές, ε, κάποια τεχνικά κοινά, τα οποία αντιμετωπίζουν και ε, ενδεχομένως προβληματίζουν όσους προσπαθούν να αξιοποιήσουν τους πόρους αυτούς. Θα θέλαμε λοιπόν να βελτιωθούν όλα αυτά και θα καταθέσουμε σχετικές ε, τροπολογίες για να καλύψουμε τα κενά αυτά προκειμένου τελικά ο κανονισμός αυτός να είναι χρήσιμος και απλός. Υπάρχει και το κείμενο το οποίο έχει ήδη εγκριθεί και διαπιστώνουμε την εισαγωγή μιας κάποιας θεσμικής ορολογίας. Για παράδειγμα, μιλάμε για το λόγο corporate, το οποίο αντικαταστά τον ε, όρο θεσμικός. Μιλάμε λοιπόν για εταιρικά συστήματα. Καλό θα ήταν λοιπόν οι νομομαθείς, ε, οι νομικοί να εξετάσουν το κείμενο. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην τα λέξει να δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για επιχειρήσεις. Όχι, πρόκειται για θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρίντσκι και θα δώσω το λόγο στην κυρία Κοσλόφσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Εκφράζω τον απόλυτο σεβασμό για τη δουλειά που κάνατε και νομίζω ότι με τις 700 και πλέον τροπολογίες που επεξεργαστήκατε καταφέρατε να ολοκληρώσετε το τιτάνιο έργο της ε, εξέβρεσης ε, συμβαστικών λύσεων. Η συνεργασία με τους κοιόδες είναι πάρα πολύ καλή και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Ως προς τα θέματα περιεχομένου τώρα, να τονίσω ορισμένα στοιχεία. Καταρχάς, το ταμείο αυτό να έχουμε υπόψη τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Ποιοι ήταν οι σκοποί του η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, της δικαιοσύνης, της συμπερίληψης, της μη διακριτικής μεταχείρισης. Σε κάθε τμήμα του Ταμείου θα πρέπει να είναι σαφείς οι και θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης πόσο ευέλικτο θα πρέπει να είναι αυτό το Ταμείο και πόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, γιατί δεν ε, ασπάζονται όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δυστυχώς τους ε, στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και υπάρχει ο κίνδυνος, ο πραγματικός κίνδυνος να μην δαπανούνται τα χρήματα, τα κονδύλια αυτά προς τον σκοπό που χορηγούνται. Η ιδέα σύνδεση λοιπόν του Ταμείου με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί μία κάποια εξασφάλιση μια δίκλυδα ασφαλεία. Ε. Και πιστεύω ότι δεν βλάπτει την ευελιξία. Υπάρχει δυνατότητα ανταπόκριση σε κάποια συγκεκριμένα περιστατικά. Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν ασφαλώ να λέμε ότι υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αντίθετο προς τον χάρτη των δικαιωμάτων, προς τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υποστηρίζω τις τροπολογίες αυτές ε, που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο υπάρχουν ε, και συστάσεις για τα κράτη-μέλη και είναι σωστό ότι επισημαίνουμε πώ μπορούν να δαπανηθούν λοιπόν τα χρήματα αυτά σύμφωνα με τις αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα λοιπόν που μας ε, απασχολεί επίσης είναι το θέμα των ελεγχών. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει σωστό έλεγχο ε, των στόχων της Ευρωπαϊκής, του, του, του Ταμείου αυτού για να πετύχουμε ακριβώς τους στόχους που έχουν τεθεί και προκειμένου να μην βρεθούμε το ταμείο αυτό να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς στόχους. Ένα παράδειγμα, το θέμα της ε, νοοτροπίας σε ό,τι αφορά το φύλλο. Μία περίεργη συζήτηση σε κάποια στην Βουλγαρία η κυβέρνηση δεν έχει προσυπογράψει, δεν έχει επικυρώσει την διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης. Γιατί, γιατί ο καθένας ενδεχομένω κατανοεί με διαφορετικό τρόπο το θέμα της ισότητας των φύλων. Αυτό αποτελεί θέμα κλειδί. Και η σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, με τις καθολικές αυτές αξίες, είναι πολύ σημαντική. Κλείνοντας, γιατί και αυτό το ταμείο, όπως και άλλα ταμεία, επηρεάζει και την κινητικότητα των νέων. Υπάρχει δραστηριότητα αυτή για τους νέους. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι ένα βασικό ζήτημα είναι η έλλειψη γνώσεων ξένων γλωσσών. Και καλό θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να εξοπλιστεί με προγράμματα. Εδώ υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των νέων. Αυτό ενδεχομένω να φαίνεται περίεργο και παρόλα αυτά ισχύει. Ευχαριστώ. Thank ε, Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Για όλες τις συνεισφορές η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης θα λάβει χώρα στις 26 με 27 Νοεμβρίου. Είναι αρκετά σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. Να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης τώρα. Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Η κυρία Μάκιντα έχει το, λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδες συζητητές για την πολύ ενεργή συμμετοχή τους. 449 ε, τροπολογίες έχουμε λάβει στο σχέδιο γνωμοδότησης. Και πριν προχωρήσω πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να, θέσω, να επιστρέψω την προσοχή των, των συναδέλφων στη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Επιτροπής Γιούρη ως ε, ε επιτροπή και ΜΟΝ. σε ό,τι φορά τι αρμοδιότητες των μεν και των δε. Ε, η Μαρίτα Ουσγκοκ από κοινού με, τον, με προεδρία, τον πρόεδρο του, της Γιούρη, τον κύριο Σβόμποντα, έγραψαν στη Σέλια Έκστρομ ως πρόεδρος της ECC ε, όπου γίνεται αναφορά στη συμφωνία στην οποία φτάσαμε. Η Επιτροπή μας ακολουθεί τον κανόνα 54 ε, σε μια σειρά από εκτιμώντας και άρθρα. Εξέτασα και τις 449 τροπολογίες και πιστεύω ότι μόλις 180 περίπου από αυτές εμπίπτουν στις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να προτείνω οι σκιώδεις συγητές να εξετάσουν μόνο τις τροπολογίες ε, που σχετίζονται με τα άρθρα και τα εκτιμώντα για τα οποία έχουμε αρμοδιότητα. Είναι σημαντικό αυτό, διότι ε, οι συντονιστές περνάνε πολύ χρόνο να υπερασπίζονται τις θέσει της Επιτροπής Απασχόλησης όταν άλλε επιτροπέ προσπαθούν να μπουν στα χωράφια μα Είναι λοιπόν λογικό όταν εμεί είμαστε η Επιτροπή συνομοδότηση, ε, ε, όταν υπάρχει μάλλον η Επιτροπή Γνωμοδότησης όπως η Επιτροπή Γιούρι, η Βασική Επιτροπή, εμεί να ακολουθήσουμε του κανόνε. Ε, δεν θα αναφερθώ βέβαια σε όλο τον κατάλογο, αλλά γιατί όχι δηλαδή κιόλα. Ε, οι τομεί όπου έχουμε αρμοδιότητα είναι τα εκτιμώντας 12, 19, 20, 27, 28, 44, 55 και 56. Και τα άρθρα είναι το 86 γ παράγραφος 3, 86 δ, σημεία J και K, όλο το 87 F, όλο το 86 L, το 86 M, παράγραφος 4, 104 α, 113, 163 ε, 168, 160 N και 160 O σημείο 4. Ε, ε, εάν θέλει κάποιος να έχει τον κατάλογο αυτόν, μπορούμε να το μοιράσουμε, να σας μοιράσουμε εν πάση την επιστολή που στείλαμε στην κυρία Βίξτρομ που αποτυπώνει τη συμφωνία μας. Προσπάθησα να είμαι ρεαλίστρια σε ό,τι αφορά το τι μπορούμε να πετύχουμε στα πλαίσια της οδηγίας αυτής. Ε, η αρχική στόχη της οδηγίας δηλαδή ε, με βάση τη αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Ε, είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε κανόνας προκύψει να είναι απλός, να είναι απλή οι κανόνες αυτοί, να είναι ενιαίοι, να είναι σαφείς, να μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και να διευκολύνουν την κινητικότητα προστατεύοντας ταυτόχρονα τους εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ των οποίων βεβαίως και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι κανόνες οι οποίοι δεν είναι σαφείς, οι οποίοι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμηνείες από χώρα σε χώρα και έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή και υπάρχει ο κίνδυνος του κατακαιρματισμού της εσωτερικής αγοράς. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε τις κατάλληλες διατάξεις έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, να περιλαμβάνονται εδώ μέτρα για την καταπολέμηση των εικονικών εταιριών ε, ό,τι και να θεσπίσουμε πάντως πρέπει να είναι λογικό, να είναι αναλογικό και οι κανόνες ε, δεν πρέπει να αποτρέπουν έναν επιχειρηματία από το να διευρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητε ε, πέρα από τα σύνορά του. Εγώ συμφωνώ με μέτρα τα οποία θέλουν να βελτιώσουν την ενημέρωση, τη διαβούλευση ε, των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους όλα αυτά στα πλαίσια μια ορθώ λειτουργούσα νομοθεσία. Εκεί που αντιμετωπίζω πρόβλημα είναι όταν γίνεται προσπάθεια να επεκτείνουμε την οδηγία αυτή και να καλύψουμε πτυχέ με τι οποίε εγώ μπορεί να συμφωνώ, αλλά δεν έχουν θέση σε αυτή την οδηγία. Η ιδέα του να καλύψουμε ε, την ποικιλομορφία, αυτό είναι κάτι που το υποστηρίζω. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την οδηγία δεν νομίζω να είναι το κατάλληλο εργαλείο. Διότι οι αναδιαρθρώσεις που μας απασχολούν εδώ έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο, στο εργατικό δυναμικό. Ε, πρέπει λοιπόν να γίνει εδώ μία ανάλυση και να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποκλίνουμε από το στόχο μας και να προσθέσουμε άλλα στοιχεία, να τα ε, στριμώξουμε εδώ με έναν τρόπο που δεν, ε, δεν φέρνει και αποτέλεσμα. Συμφωνώ βεβαίως με επιμέρους μέτρα που έχουν να κάνουν με τις εταιρείε που προσπαθούν να παραβιάσουν την νομοθεσία, τις εικονικές εταιρείε, ε, πρέπει να οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι γι' αυτό και σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις ε, διαχείρισης και τις ε, διάφορες αναφορές για τις ζητηνακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Θέλουμε ε, πιο απλούς κανόνες για την ε, συμμετοχή, την εμπλοκή των εργαζομένων. Είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι τροπολογίες. Θα ετοιμάσω συμβαστικές προτάσεις, θα τις στείλω και όλους πριν από την πρώτη συνάντησή μας που θα λάβει η χώρα στις 25 του μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Μάκιντάιρ. Δεν θέλω να ξεκινήσω τώρα μια νέα συζήτηση, απλώς να πω ότι η Γιούρη είναι η επιτροπή που ηγείται εδώ για αυτήν την έκθεση σχετικά με τις συνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Εμείς ε, είμαστε συνδεδεμένοι ε, επικουρική επιτροπή με βάση το άρθρο 54 με μικτές ε, αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη συμμετοχή των εργαζομένων, καθώ και μια σειρά από εκτιμώντα τα οποία αναφερθήκατε νωρίτερα. Ε, και έχουμε συνηθίσει να συνεργαζόμαστε με άλλε επιτροπέ. Προφανώ και θα φροντίσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά εμεί θα μιλήσουμε για τι θέσει τη Επιτροπή Απασχόληση, για ζητήματα που αφορούν την απασχόληση. Ε, και θα κάνουμε βεβαίω ε, ό,τι περνάει από το χέρι μα για να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί και πέρα ε, θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδους εισηγητές. Ο κύριος Σόγκορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ με την εισηγήτρια να περιοριστούμε σε αυτά που είναι των αρμοδιοτήτων μας. Θα θέλω να περιορίσω τα σχόλιά μου σε ένα-δύο ζητήματα αρχής. Γενικότερα θέλω να επαναλάβω αυτό που είπατε κατά την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης Εάν, εάν θέλουμε οι επιχειρήσεις να επιχειρήσουν ελεύθερα στην ενιαία αγορά, χρειαζόμαστε σαφείς, απλούς και εύκολα εφαρμόσιμους κανόνες. Καλωσορίζουμε τις τροπολογίες που πάνε προς την κατεύθυνση του να δώσουν στις επιχειρήσεις να συνδυάσουν τις εκθέσεις προς τους μετόχους και προς τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι σαφείς πληροφορίες στις εκθέσεις αυτές και περιορισμένες μόνο σε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα. Σε ό,τι αφορά την, τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης, πολλές τροπολογίες εδώ δημιουργούν διπλούς κανόνες, διότι εκεί έχουμε ήδη κανόνες ευρωπαϊκούς ε, που λειτουργούν ε, στην οδηγία 14 του 2002 δεν νομίζω να χρειάζεται εδώ να υπάρξει σύγχυση ή και επικάλυψη Αναμένουμε ανυπομονησία τη συζητήση για να βρούμε τι σωστέ λύσει ό,τι αφορά τα δικαιώματα συμμετοχή των εργαζομένων. Να πω όμω αυτή τη αρχή ότι το κανόνα των 10 ετών που προτείνουν κάποιοι για την έγκριση νέων κανόνων μας, μου φαίνεται υπερβολικό. Αναμένω να έχουμε μια καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και του συνεισηγητέ και του συνεισηγητέ του και Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μίκαλ Ντέτχεν έχει τώρα το λόγο για τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμη συνάδελφοι. Οι δικέ μου αξιώσεις είναι πολύ απλές. Οι, οι εργαζόμενοι έχουν ε, τα ίδια δικαιώματα όπως και οι επιχειρήσεις. Ο πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ισορροπημένη. Η οικονομική Ευρώπη θα πρέπει να είναι και κοινωνική Ευρώπη και να προχωρήσει και κοινωνικά. Ιδάλλως θα χάσουμε την ισορροπία μας και θα χάσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Καλό θα ήταν ε, αν οι εργαζόμενοι μπορούσαν να έχουν το δικαίωμα αυτό και να το μεταφέρουν αυτό το δικαίωμα από εργοδότη σε εργοδότη. Αυτό δεν ισχύει στην παρούσα φάση. Οι εργαζόμενοι Στη Γερμανία, για παράδειγμα, πρέπει να αποδεικνύουν διάφορα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή του σε μετοχικέ εταιρείε. Αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό λοιπόν η ομάδα μου και εγώ ζητάμε μια οριζόντια δίγεια για το δικαίωμα των ε, εργαζομένων. Μια οδηγία πλαίσιο για την ε, συναπόφαση και για την αυτονομία των τιμών το καλύτερο θα ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είχε νέα ελάχιστα πρότυπα ε, για τους εργαζόμενους μέσω της ε, συναπόφασης ε, μέσω διοικητικών συμβουλίων. Αυτό που συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα φάση για την προστασία των εργαζομένων είναι δύσκολο, περίπλοκο και αδιαφανές. Και γι' αυτό λοιπόν έχω καταθέσει σχετικέ τροπολογίε. Χρειαζόμαστε απλούς κανόνε, εφικτού και πραγματική προστασία για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ε, μια ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας εγκατάστασης στην κρατημέλη και το δικαίωμα προστασίας. Το δικαίωμα εγκατάστασης, αυτή η ελευθερία εγκατάστασης θα πρέπει να συνδεθεί με μια σχετική κοινωνική ευθύνη και η επικουρική προστασία των δικαιωμάτων αυτών δεν μπορεί να έρθει με την οδηγία αυτή. Χρειαζόμαστε προστασία επίσης του δικαιώματος συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση των επιχειρήσεων για 10 τουλάχιστον χρόνια προκειμένου να μην δημιουργούνται κίνητρα για μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων που θα έχει ως μοναδικό στόχο την αποφυγή της συνδιαχείρισης από πλευρά των εργαζομένων. Και εγώ και οι συναδελφοί μου ελπίζουμε να είναι επικοδομητική συνεργασία, η επικουρικότητα δεν αποτελεί μόνο ένα θέμα το οποίο αναφέρουμε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Και χρειαζόμαστε λοιπόν σαφείς και ξεκάθαρες εγγύησεις για τους εργαζομένους και θα ήθελα τέλος να ζητήσω μεγαλύτερη κοινωνική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ε, Ευχαριστούμε κύριο Σελίμοβιτς. Um, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με την εισηγήτρια να συγκεντρωθούμε στα σημεία εκείνα που μας απασχολούν, εμάς δηλαδή, προς αρμοδιότητάς μας. Ε, ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Αλλά θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο η γενικότερη εντύπωση που υπάρχει για αυτή την έκθεση, για μένα τουλάχιστον, είναι κάπως, ε, με κάνει κάπως διστακτικό. Την υποστηρίζουμε, αλλά η συγχώνευση, η μετακίνηση των επιχειρήσεων θεωρείται τελικά ως κάτι αρνητικό. Αυτή είναι η εντύπωση που δίνεται, ότι είναι ίσως επικίνδυνο, ότι εγώ, εγώ δεν συμφωνώ όχι επειδή η ελεύθερη μεταφορά και των επιχειρήσεων είναι βασικό στοιχείο της συνθήκης, αλλά και επειδή αυτή είναι η απάντηση στα προβλήματα που έχουμε. Εάν θέλουμε να βελτιώσουμε ε, τους ρυθμούς ανάπτυξης, ε, να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν και νέες θέσεις απασχόλησης, τότε όλα αυτά, η διάσπαση, οι συγχωνεύσεις, ε, πρέπει να ενθαρρυνθούν και κατ' εμέ η έκθεση ε, θυμίζει λίγο αυτόν τον, ε, τον, τον, αυτό το δισταγμό και αυτόν τον σκεπτικισμό απέναντι σε αυτή την ελευθερία. Και πρέπει να το πω. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση, πρώτα απ' όλα εμείς πιστεύουμε, προτείνουμε τη δημιουργία μίας έκθεσης ε, έτσι ώστε να αποφύγουμε το διοικητικό άχθος. Να πω όμως εδώ και το εξής έχουμε διαφορετικές παραδόσεις στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Στη Νότια Ευρώπη οι εργοδότες είναι απέναντι στα συνδικάτα. Στη Βόρεια Ευρώπη όμως συνεργάζονται. Mm. Έχω την εντύπωση ότι τους τελευταίους μήνες οι εκθέσεις αυτής της Επιτροπής έτσι τίνουν προς το νότιο μοντέλο. Προσπαθούμε στην νομοθεσία να πούμε ποια είναι τα δικαιώματα των εργοδοτών, ποια των εργαζομένων και δίνουμε μια μάχη. Όχι, εμείς δεν εργαζόμαστε έτσι. Θεωρούμε ότι έτσι καταστρέφουμε το βόρειο μοντέλο, το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά. Συνεργαζόμαστε με τα συνδικάτα, οι εργοδότες και τα συνδικάτα ε, τα βρίσκουν. Δεν, δεν παρεμβαίνει το κράτος. Υπάρχει απόλυτη αυτονομία. Και θα ήθελα να το πω και στα πλαίσιο της έκθεσης αυτή. Θα θέλαμε η έκθεση αυτή να εξεταστεί αυτόνομα από τους εργοδότες και τους εργοζόμενους Έχουν τρόπο να το κάνουν. Ε, το κράτος ε, δεν έχει δουλειά εδώ να εμπλακεί Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μόνο μία έκθεση, αλλά θα πρέπει να γίνει σεβαστή αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Τώρα, η τροπολογία 50, εδώ υπάρχει ορισμός των τεχνητών συμφωνιών. Ε, σημαντικό, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτές οι τεχνικές συμφωνίες ε, ορίζονται τελώς διαφορετικά από χώρα σε χώρα της Ένωσης. Δεν θα ήθελα λοιπόν να ε, χαμηλώσουμε τα πρότυπα που έχουμε εμείς λόγω κάποιων άλλων. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη να είναι αυτά που θα αποφασίσουν ποια θα είναι αυτά τα πρότυπα. Ιδάλω ε, θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε ένα κοινό επίπεδο και θα είναι προ τα κάτω αυτή η εξίσωση. Πολλέ χώρε θα πρέπει να δεχθούν δηλαδή ε, να, ε, να, να χαμηλώσει το επίπεδο των προδιαγραφών για το τι είναι τεχνητή συμφωνία έχουμε υποβάλει μια πρόταση να έχουμε αντικειμενικούς ε, λόγους ε, για, την, τον των τεχνητών συμφωνιών, ε, τεχνητών διακανονισμών. Ε, είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει επίσης και ο όρος adequate προς appropriate payments, ότι αφορά τις πληρωμές δηλαδή. Ε, λέμε ότι πρέπει να είναι κατάλληλο, διότι ορισμένε φορές το κράτος αγοράζει μετοχές, γιατί γνωρίζει, έχει πληροφορίες που δεν έχει ε, ο μέτοχος. Ε, και το κράτος ε, κάνει μια πρόταση που είναι υποχρεωμένο να δεχτεί η επιχείρηση. Το appropriate είναι κάτι άλλο. Οι μειοψηφόντες με μετοχή πρέπει να έχουν προστασία και πρέπει να έχουν και τις πληροφορίες που έχουν οι υπόλοιποι. Τώρα, ο, διάβασα το άρθρο 86 και το μηχανισμό προσφυγών. Ε, εντάξει, αλλά τα κράτη-μέλη που δεν είναι υποχ... ε, ε ικανοποιημένα με το επίπεδο θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν ε, να μπορούν να προσφύγουν στο Εθνικό Δικαστήριο εφόσον δεν συμφωνούν. Αναμένω τις συζητήσεις του και του συζητητέ. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ε, έτσι ώστε να αντιληφθούμε ότι η κινητικότητα των επιχειρήσεων ε, στην Ευρώπη είναι μία λύση στα προβλήματά μας και όχι ένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σελίμοβιτς. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόμπος Πελμέρια, δεν είναι εδώ όμως και δεν έχει δώσει αντικαταστάτη. Επίσης εκπρόσωπος των Πρασίνων δεν είναι εδώ και δεν έχει ορίσει αντικαταστάτη. Αυτό σημαίνει ότι ακούσαμε ε, όλους όσοι είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Φαίνεται ότι θα κάνετε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ε, κυρία ε, Μακεντάιρ, αν θέλετε σας ξαναδίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ ε, όλους. Ε, πραγματικά πρέπει να συναντηθούμε. Προσδοκώ αυτές τις συναντήσεις ε, και τις αναμένω λοιπόν με τις συναντήσεις με τους Κιώδης έτσι ώστε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά. Και είμαι βεβαία λέει η Πρόεδρος ότι θα έχετε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και συνεργασία. Εξέταση τροπολογιών σήμερα 18 Οκτωβρίου. Έγκριση ε, στην ΕΜΠΛ 15 Νοεμβρίου και στην Euro στις 20-21 Νοεμβρίου. Η επόμενη συνεδρίαση να σας υπενθυμίσω σχετικά με το θέμα αυτό ότι η επόμενη συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για την 5η Νοεμβρίου έχει ακυρωθεί και επομένως η επόμενη συνεδρία θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο και μετά άλλη μία στις 19 Νοεμβρίου και στις 20 Νοεμβρίου ε, στις Βρυξέλλες. Επομένως θα έχουμε πολλές μαζεμένες συνεδριάσεις σε τέλη ε, Νοεμβρίου, αλλά η συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου έχει ακυρωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ ε, που είστε εδώ. Η Πρόεδρος ευχαριστεί τους Γερμινείς, ευχαριστούμε και εμείς. Και πραγματικά δεν τα κατάφερα να ε, πω στους ε, ομιλητές που πήγαιναν πολύ γρήγορα να ρυθμίσουν λίγο το ρυθμό τους, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα κάνω καλύτερα την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε, χαίρετε.